Sir Robert, can we start? Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Sir Robert, χρειαζόμαστε την άδειά για να αρχίσουμε. Επίτες το λέγεται συνήθως με προλαβαίνει. Αυτή τη φορά ήθελα να το προλάβω εγώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην Επιτροπή μας τον κύριο Κρίστιαν Λέφλερ, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΕΔ για τη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Θα μας ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων ε, σε ό,τι αφορά το διάλογο και τη συμφωνία συνεργασίας με την Κούβα, αλλά θα μας ενημερώσει και για τις υπόλοιπες εξελίξεις στη Λατινική Αμερική. Έχετε το λόγο. Ελπίζω να είναι για σας ε, ευχάριστο και απολαυστικό. Η τιμή είναι δική μου. Θα ήθελα μια σύντομη ενημέρωση καταρχήν ε, για την πορεία των διαδικασιών σε ό,τι αφορά την έναρξη, την εδραίωση ή την αναβάθμιση των ε, συμβατικών μας σχέσεων ενοχικό, είναι σημαντικό μας σχέσιο με τη Λατινική Αμερική. Ο νέος στην παρέα μας, το νέο και τον The Block, θυμάστε την, το συγκρότημα αυτό, είναι η Κούβα. Πρόσφατα το Συμβούλιο έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΙΕΔ εντολή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για έναρξη πολιτικού διαλόγου και συμφωνία συνεργασίας με την Κούβα. Και αυτό ήταν το αντικείμενο αρκετά σφοδρών συζητήσεων και μακροχρόνιου προβληματισμού των κρατών μελών πριν αποφασίσουν να δώσουν τελικά αυτή την διαπραγματευτική εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕΔ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στόχος αυτών των ε, κατευθυντηρίων γραμμών και της διαπραγματευτικής εντολής για σύναψη συμφωνίας με την Κούβα, όπως προβλέπει αυτή η διαπραγματευτική εντολή, δεν είναι να αλλάξει άρδεν η πολιτική μας απέναντι στην Κούβα. Η διαπραγματευτική αυτή εντολή εξασφαλίζει συνέχεια της υλοποίησης των στόχων και μία επίσης συνέχεια της προσέγγισης μας. Ο πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, ε, στη σχέση με την Κούβα είναι γνωστός εδώ και πολύ καιρό. Στόχος μας είναι πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε και τον εξυγχρονισμό της Κούβας, να ενθαρρύνουμε για μεταρρυθμίσεις και να διευρύνουμε το πεδίο των κουβανών για άσκηση των ε, δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Αυτός ήταν γνωστός, δεδηλωμένος και αμετάβλητος ε, ανέκαθεν στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό προβλέπει και η διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου και θα είναι και ο στόχος της ε, μελλοντική μας συμφωνίας με την Κούβα. Τι έχει αλλάξει λοιπόν, αν ο στόχος είναι ο ίδιος. η αλλαγή οφείλεται στις εξελίξεις, στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Κούβα. Οι εξελίξεις είναι αργές, αλλά σταθερές. Χρειάζεται μεγάλη εξουδέρκεια και η όβια υπομονή για να παρακολουθήσει κανείς και να εντοπίσει, να αντιληφθεί αυτές τις αμυδρές αλλαγές που γίνονται στην Κούβα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αλλαγές και μερικές μάλιστα είναι και σημαντικές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την οικονομία, τις κοινωνικές δομές και σε κάποιο βαθμό αφορούν και την ουσία της πολιτικής και των πολιτικών δικαιωμάτων. Είναι γνωστό τη σπάση, αλλά είναι γνωστό και στους κουβανούς ότι θα θέλαμε η διαδικασία αυτή να προχωρήσει ταχύτερα και θεαμα... θεαματικότερα. Το θέμα είναι όμως πώς θα συμπαρασταθούμε σε αυτή τη διαδικασία και αυτός είναι ο στόχος της συμφωνίας. Η συμφωνία μας εξασφαλίζει ένα πλαίσιο, θα έλεγα και ισχυρό πλαίσιο, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καν συμβατικό πλαίσιο, γιατί δεν έχει συναυθεί ακόμη αυτή η συμφωνία. Πάντως, εφόσον συναυθεί, η συμφωνία θα μας εξασφαλίσει ένα πλαίσιο για πολιτικό διάλογο και συνεργασία, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος μας και να στηρίξουμε τις αλλαγές στην Κούβα, να βοηθήσουμε για μεγαλύτερη, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη συμμετοχή και μεγαλύτερο δυναμισμό στην Κούβα προς το συμφέρον και το όφελος των κουβανών πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει συνεργασία με την Κούβα και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό για 25 ολόκληρα χρόνια. είχαμε μια διακοπή στη συνεργασία μας, τελευταία 20, 25 ετία, αλλά το 2008 την ε, επαναλάβαμε. Και ελπίζω να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία και να είναι πιο εστιασμένη. Έχουμε και διάλογο με την Κούβα. Πολιτικός διάλογος υψηλού επίπεδου, όχι πολυτακτικός, αλλά τακτικός ήταν ο τεχνικός διάλογος σε επίπεδο αξιωματούχων ε, υψηλόβαθμων για τεχνικά θέματα όπως η γεωργία, οι κλιματικές αλλαγές, πρόληψη θεομηνιών, φυσικών καταστροφών και διάλογος ακόμη και για κάποια πολιτικά θέματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε και αυτόν τον διάλογο να τον ενισχύσουμε και να το εξασφαλίσουμε μία ισχυρότερη βάση. Αλλά όπως βλέπετε είχαμε διάλογο σε πολλά επίπεδα, πολιτικό, κοινωνικό, τεχνικό και αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο ενημερωμένοι και να έχουμε πιο εμπεριστατωμένη γνώση για τη συνέχεια του διαλόγου αυτού. Έχουμε λοιπόν τις ε, κατευθυντήριες εντολές του Συμβουλίου που διαμορφώνουν τη διαπραγματευτική μας εντολή. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σα αφήσει εδώ και πολλά χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών αυτών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν και πολύ συνεπής. Πάνω από τις μισές χώρες μέλη μέχρι στιγμής έχουν συνάψει τις δικές τους συμφωνίες, μνημόνια συνεννόησης, δηλώσεις, διακηρύξεις με την Κούβα και έχουν ξεκινήσει διάλογο και συνεργασία διμερή. Μερικές φορές ο διάλογος αυτός και η συνεργασία συνάδουν με την κοινή προσέγγιση θέση και πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μερικές φορές τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες δεν έχουν πολύ άρρηκτο δεσμό μαζί τους. Οπότε ελπίζουμε ότι θα έχουμε ελπίζουμε ότι σε μια κοινή προσέγγιση σε ένα κοινό διάβημα ή εγχείρημα θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια πιο κοινή προσέγγιση και ένα κοινό όραμα σε ό,τι αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κούβα. Και αυτό θα είναι προς όλων μας και κυρίως προς όφελος της Κούβας και των πολιτών της. Είναι σημαντικό να έχουμε μια πιο περιεκτική και πιο καθιερωμένη και δρεωμένη προσέγγιση. Έχουμε λάβει λοιπόν τις διαπραγματευτικές εντολές και την απόφαση για τις ε, διαπραγματευτικές εντολές του Συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου. Τις ε, διαβιβάσαμε στην ε, κοβανική κυβέρνηση λέγοντας ότι έχουμε πλέον εξουσιοδότηση για έναρξη της διαπραγμάτευσης. Και έχουμε λάβει και επίσημα την απάντηση της κουβανικής κυβέρνησης ε, με έκφραση ενδιαφέροντος ε, για την ένδειξη των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις γιατί δεν τα βρήκαμε ακόμη στο χρονοδιάγραμμα, δεν βρήκαμε κατάλληλες ε, και συμβατές ημερομηνίε. Ψάχνουμε όμως την κατάλληλη στιγμή που θα συμπέσουν τα προγραμματά μας και θα μπορέσουμε και εμείς και οι ομόλογοι μας στην Κούβα να βρούμε μια στιγμή τον κατάλληλο χρόνο για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια και να αρχίσουμε να χαράζουμε το δρόμο προς μια συμφωνία. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, εν συντομία κύριε Πρόεδρε, θα σας πω πώς έχουν άλλες εκρεμείς διαδικασίες. Αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Στις 21 Μαρτίου θα έχουμε στις Βρυξέλλες συνεδρίαση των επικεφαλής ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων της Μερκοσούρ. Οπότε και ο αρμόδιος της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Μασάντο, θα λάβει μέρος για να δούμε σε τι φάση της διαδικασίας απελευθέρωσης βρισκόμαστε. Αν κρίνουμε τη διαδικασία αυτή ικανοποιητική θα μπορέσουμε να δώσουμε νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο προκειμένου να καταλήξουμε σε ε, ε, διεκπαιρέωση των διαπραγματεύσεων και μάλιστα στο εγγύς μέλλον. Μέχρι στιγμής είχαμε αρκετές δυσκολίες, κυρίως ε, στις χώρες Μερκοσούρ. Δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει τι μορφή θα δώσουν στην προσφορά του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακούσει φημολογίε για το τι χαρακτηριστικά θα έχει, αλλά ακόμη την περιμένουμε αυτή την ενιαία προσφορά από τη Μαρκοσούρ. Και ευελπιστούμε ότι θα είναι αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσφορά για να την κρίνουμε ω ικανοποιητική βάση και να περάσουμε στον τελικό γύρο των διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι τόσο ικανοποιητική αυτή η προσφορά. Πάντως πιστεύω ότι μετά τη συνεδρίαση στο τέλος εβδομάδας, οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου θα σας ε, ενημερώσουν για τις προπτικές που ανοίγει ή όχι αυτή η συνεδρίαση. Πάντως, εμείς είμαστε πρόθυμοι ε, για ενεργό συμμετοχή προκειμένου να προωθήσουμε τη συμφωνία. Τώρα, για μη εμπορικά θέματα, ε, για τις συμφωνίες σύνδεσης και κυρίω στο σκέλο αναπτυξιακή συνεργασία. Εκεί έχουμε κάποιε εκκρεμότητε, αλλά είναι ίσονα σημασία σε σχέση με τι προκλήσει ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τι εκκρεμότητε που έχουμε σε οικονομικά και εμπορικά θέματα. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στο Εκουαδόρ δεύτερος επίσημος γύρος διαπραγματεύσεων για να ενταχθεί και το Εκουαδόρ στην πολυμερή Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κολομβία και το Περού. Είχαμε τον πρώτο επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων τον Ιανουάριο, μετά από σωρία προπαρασκευαστικών ε, συνεδριάσεων το πρώτο εξάμεινο του προηγούμενου έτους. Η κατάσταση είναι πολλά υποσχόμενη γιατί φαίνεται ότι το Εκουαδόρ είναι προσιλωμένο στην, ε, στο στόχο αυτό και έχει επίγνωση τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το κοινό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν ήδη η Κολομβία και το Περού. Βέβαια οι προκλήσεις είναι μεγάλες γιατί το Εκουαδόρ μας έχει επισημάνει πολλούς τομείς για τους οποίους θεωρεί ότι χρήζει ιδιαίτερη μεταχείρισης εξαιτία των κοινωνικών οικονομικών διαφορών που παρουσιάζει σε σχέση με την Κολομβία και το Περού. Επίσης, ανέκυψαν και νέα εμπορικά θέματα, θέματα μη δοσμολογικών φραγμών στο εμπόριο. Είναι νέα στοιχεία που ανέκυψαν τους τελευταίους μήνες και που επιβραδύνουν κάπως το ρυθμό των διαπραγματεύσεων, που ελπίζαμε να είναι πιο γοργός. Πάντως θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση και αυτό το δεύτερο επίσημο γύρο των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στο Κίτο. Τώρα, στα άλλα δύο πλαίσια προσπαθούμε να κάνουμε μια αναβάθμιση των σχέσεών μας για το Μεξικό και τη Χιλή. Με το Μεξικό Δημιουργήσαμε μια κοινή ομάδα εργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό για να δούμε τους τρεις ε, πυλώνες της εργασίας ε, για το θέμα αυτό. Είχαμε και μια κοινή συνάντηση που προβλέπεται μέσα Φεβρουαρίου στο Μεξικό και έχουμε σημειώσει πρόοδο για να ορίσουμε ένα κοινό όραμα για το πώς θα μπορούσε να δημορφωθεί μια μελλοντική αναβαθμισμένη συμφωνία. Θα γίνουν περαιτέρω ανταλλαγέ τους επόμενους μήνες και πιο πολλές θα είναι εικόνικες μέσω τηλεδιάσκεψης ενδεχομένω και μια κατηδίαν συνάντηση αργότερα μέσα στην Άνοιξη με σκοπό να οριστικοποιηθεί μια κοινή έκθεση τμήματο, σε ό,τι αφορά ε, την ε, ανάληψη των εργασιών το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια του θερινών διακοπών σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή της αναβάθμιση αυτή των σχέσεων και εμείς και οι Μεξικανοί θεωρούν ότι θα είναι φιλόδοξοι αυτή η ανεβάθμιση. Θα γνωρίζετε ότι οι Μεξικανοί ήθελαν να ενοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις πέρσι με την Αμερική, με το TTIP. Αλλά ούτε εμείς, ούτε οι Αμερικανοί δεν θέλαμε να είναι πολυμερείς αυτές οι διαπραγματεύσεις. Επίσης, το Μεξικό αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται να ολοκληρώσουμε την διαπραγματεύση ε, ΣΥΤΑ και SPA. Και ενώ αυτές οι καθολικές συμφωνίες έχουν συνδραματίσει σημαντικό ρόλο τα τελευταία 12 χρόνια, ε, εν ώψη και των σχέσεων ε, μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, καταλαβαίνουμε ότι έχει έρθει η χρονική στιγμή να είμαστε πιο φιλόδοξοι και στη σχέση μας με το Μεξικό. Και είμαστε αισιόδοξη ότι αυτή η έκθεση οράματος θα αποτυπώσει αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας προκειμένου και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου να καταθέσουν μια σχετική πρόταση γιατί πρέπει να γίνουν διάφορα προπαρασκευαστικά βήματα, μελέτη αντικτύπου και το καθεξής, αλλά να δοθεί εντολή τελικά τέλη του έτους και αρχές ε, του επόμενου έτους. Με τη χειλή είμαστε λίγο, έχουμε μείνει λίγο πίσω συμφωνήσαμε ότι επί της αρχής θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την ε, Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής και πριν από κάποιες μήνες προσφάτως λάβαμε σχετικές προτάσεις από τη Χιλή για το επίπεδο της αναβάθμισης ε, είναι κάπως πιο χαμηλές από τις προσδοκίες μας και διεξάγουμε μια συζήτηση με τις αρχές της Χιλής στην παρούσα φάση για να διευκρινίσουμε κατά πόσο μπορούμε να αυξήσουμε τον πύχη των φιλοδοξιών προκειμένου να φτάσουμε πιο κοντά στο δικό μας όραμα και να μην απέχουμε υπερβολικά από αυτό που φανταζόμαστε και στο Μεξικό, για το Μεξικό. Και αυτό θα συμφωνούσε με την ε, αρχή ότι θέλουμε επίπεδο παρόμοιο φιλοδοξίας ε, με τους τέσσερις εταίρους μας στην περιοχή του Ειρηνικού, γιατί έχουμε τέτοιες ε, τέτοιο επίπεδο με το Περού, για παράδειγμα. Θέλουμε αντίστοιχο επίπεδο και με τη Χιλή και με την Κούβα. Θα θέλαμε λοιπόν να συζητήσουμε για να δούμε και να δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση και με τη χειλή. Δεν ξέρω πρόεδρε, μάλλον μακρηγόρησα, θα ζητώ συγγνώμη, αλλά ήθελα να σας παρουσιάσω την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σολαφράγκα. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Λέφλερ που ήρθε και μας έκανε μια γενική επισκόπηση της κατάστασης για τις σχέσεις μας με τις χώρες της ε, Νότιας κυρίως Αμερικής. Ε, είναι σημαντική μια τέτοια συζήτηση και πολύ επίκαιρη, γιατί έχουμε προσανατολισμό που θα πρέπει να τον κρατήσουμε και να μείνουμε προσιλωμένοι στη, στο θέμα αυτό της αναβάθμισης των σχέσεών μας με τη Λατινική Αμερική. Ε, θα ξεκινήσω το σχόλιο μου με την Κούβα. Μας είπατε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών οφείλεται στις αλλαγές ε, στην πολιτική της Κούβας και η νέα διαπραγματευτική εντολή. Το γεγονό ότι δόθηκαν διαπραγματευτικέ εντολέ για την σύνευση συμφωνία για πολιτικό διάλογο και συνεργασία σηματοδοτούν ε, σημαντική αλλαγή, γιατί η Κούβα είναι η μοναδική χώρα τη Λατινική Αμερική που δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνδέεται με καμία, κανένα τρόπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε το, το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πόσο προσιλωμένοι είμαστε σε αυτό, τα βραβεία Ζαχάροφ που δίνουμε τα τελευταία χρόνια και δεν θα πρέπει ε, η ανομαλία αυτή σχέση με την Κούβα να αποδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα διαπιστώσετε και στην ΕΕΔ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποτέ δεν έθεσε προσκόμματα σε ό,τι αφορά την ανάθεση αυτής της διαπραγματευτικής εντολής. Και πραγματικά ελπίζουμε να είναι απτές ε, οι αλλαγές στην πολιτική της ε, Κούβας, ώστε άνθρωποι όπως ο Λουίς να μπορούν ελεύθερα να μεταβαίνουν στην Κούβα. Ερωτώ λοιπόν ε, τον κύριο Λέφλερ. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε. Ποιος ε, κατά τις προβλέψεις σας είναι ο χρονικός ορίζοντας για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας συνεργασίας με την Κούβα. Γιατί Έχουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου και ξέρουμε ότι εφόσον τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε την επιθυμία του ΕΚΟΔΟΡ να ενταχθεί σε αυτή την πολυμερή συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Και ευελπιστούμε ότι θα ευοδοθούν οι ο δεύτερος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να επιστήσετε ε, στις αρχές ε, του Εκουαδόρ την ανάγκη να, να εξασφαλίσουν μια ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις ε, γιατί ενδιαφέρονται πολλοί ευρωπαϊκέ επιχειρήσει γι' αυτό. Είναι σημαντικό θέμα να το επισημάνουμε. Τώρα, διαπραγματεύσει με το Μαρκοσούρ. Είμαι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμφωνία αυτή σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρκοσούρ. Και ήταν ιδιαίτερα εκνευριστική αυτή η κατάσταση και απογοητευτική γιατί από το 2004 είχαμε διαπιστώσει αυτή την αποτελμάτωση. Ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε μια απεμπλοκή της κατάστασης και θα συνάψουμε αυτή την ε, τεράστια σημασία συμφωνία με τη Μερκοσούρ, γιατί και η Μερκοσούρ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη πληθυσμού και από άποψη ε, ακαθάριστο χώριο προϊόντος έχουν τεράστια σημασία. Ελπίζω λοιπόν στις 21 Μαρτίου, μέχρι τις 21 Μαρτίου να υποβάλουν οι χώρες του Μερκοσούρ μια ικανοποιητική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόταση. Τώρα σε ό,τι αφορά της, την ανέωση της συμφωνίας με το, με το Μεξικό συγγνώμη, και τη Χιλή. Γνωρίζετε τη θέση μας και γνωρίζετε τη σύνοδο κορυφής με τη Σελάκ πέρυσι δώσαμε εντολή στις ομάδες εργασίας για να εντοπιστούν οι τομείς και τα κεφάλαια στα οποία θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στο μέλλον στις συμφωνίες αυτές. Στο Μεξικό έγινε μια πολύ σημαντική συνταγματική αναθεώρηση με αποτέλεσμα να ανοίξει σημαντικός τομέας του ανταγωνισμού από το άνοιγμα από το οποίο θα επωφεληθούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως ε, η απελευθέρωση στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών θα είναι πολύ επωφελής για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εδώ και πολύ καιρό ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε, αλλά επιτέλους συζητούμε τη Λατινική Αμερική. Επιτρέψτε μου να μπορέσω με κάποια άνεση χρόνου να παρουσιάσω τις απόψεις μου, γιατί δεν έχουμε πολλούς βουλευτές και θα ήθελα να μεταβάσω τον κύριο Λεφιλέρ τη θέση της ομάδας. Τώρα, ε, ξέρετε τη μεγάλη προτεραιότητα δίδουμε στις ε, ε, σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μεγάλη προτεραιότητα είναι η σύναψη της συμφωνίας και με το Μεξικό, γιατί έχει παρατραβήξει αυτό το θέμα χρονικά και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έχει επικεντρώσει όλους τους πόρους και τις προσπάθειες και την ενέργεια στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε και άλλες πολύ σημαντικές προτεραιότητες ε, όπως είναι η συμφωνία με το Μεξικό, η συμφωνία με τη Χιλή, που θα ευνοήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το ίδιο σκήκε για τη συμφωνία με τη Χιλή. Και παρακαλώ πείτε μας για τα χρονοδιαγράμματα, γιατί ο χρόνος για την πολιτική είναι πολύ σημαντικός. Ο κύριος Γιάννης είναι ο επόμενος ομιλητής. Θα σας θέλω να παρακαλούσα να μην ξεπεράσετε τα τρία λεπτά γιατί θα πρέπει να δώσουμε χρόνο και στον καλεσμένο μας να απαντήσει, να μην εξαντλήσουμε όλο το χρόνο σε ερωτήσεις. Για να επιτρέψω και στους 20 συναδέλφους που έχουν εγγραφεί στο κατάλογο μιλητών να λάβουν το λόγο, θα είμαι πολύ λακωνικός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Λεφλέρ για την παρουσία του και για τις εξηγήσεις που μας έδωσαν. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικά αυτά εδώ και 40 χρόνια με εντυπωσιάζει η διπλωματική γλώσσα που είναι πολύ κομψή αλλά δεν έχει περιεχόμενο και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό και αυτής της συνάντησης. Γιατί περισσότερο συμβολική αξία είχε η παρουσία του κ. Λεφλέρ. Ουσιαστικά πράγματα δεν ακούσαμε. Απλώς σημειώνουμε ότι δεν έγινε τίποτα σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλαφράγκα που αναφέρθηκε σε μένα γιατί γνωρίζουμε όλοι οι παρόντες και το γνωρίζει με το παραπάνω ο κύριος Λεφλέρ ότι κηρύχθηκα ε, ότι με παράνομο και πολύ αγενή τρόπο ε, εκδιώχθηκα από την ε, Κούβα παρόλο που είχα κανονική θεώρηση διαβατηρίου. Με απέπεψαν όμως. Θα ήθελα να ζητήσετε τις κουβανικές αρχές να μου επιστρέψουν ε, τα χρήματα που έδωσα για να μου δώσουν τη θεώρηση. Γιατί κάποιοι κλέφτες ε, εισέπραξαν ε, τα χρήματα που κατέθεσα για την θεώρηση του διαβατηρίου. Θα πρέπει να το επισημάνετε αυτό στις κουβανικές αρχές στις επόμενες συναντήσεις Πάντως θα ήθελα να πω ότι ούτε εσείς οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα μπορούν ε, να εκδιώκονται από την Κούβα. Θα πρέπει να μας διαβεβαιώσουν οι κουβανικές αρχές ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε στην Κούβα ελεύθερα και κάθε φορά που θέλουμε και δεν θα μας παρακολουθεί συνέχεια η μυστική αστυνομία. Και πραγματικά ε, ήταν το άκρο να αυτή η αποπομπή, όχι επειδή έγινε για μένα θα έλεγα το ίδιο αν ε, αποπεμπόταν οποιοδήποτε βουλευτής ή μέλος της Επιτροπής. Είναι πραγματικά παράδεκτη αυτή η μελος επιτροπης ειναι πραγματικα Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ, γιατί είναι γνωστές ε, οι διαστάσεις της Μερκοσούρ και η σημασία που έχει η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας. Το Μάρτιο του 2014 Προ το τέλο τη κοινοβουλευτική θητεία, ε, είναι κρίμα να μην έχουμε έστω και τυπικά μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την ανταλλαγή των προσφορών των συμβαλωμένων μερών. Είναι πραγματικά παράδεκτο. Το να μην έχουμε στοιχεία, εντάξει, αλλά το να μην έχετε συμφωνήσει οι δύο πλευρές για να χαρακτηρίσετε τόσο αποτυχημένη τη διαδικασία, τι να σας πω. Πάντως, εγώ, όπως και οι υπόλοιποι παρόντες, είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διεκπαιρέωσης των διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας σύνδεσης με το στρατηγικό εταίρο μας που είναι η Μερκοσούρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Στάνοκ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, Τα αγγλικά σας είναι τέλεια που δεν ξέρω αν έρχεστε κι εσείς από την χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα από όλε. Σε κάθε περίπτωση όμως συγχαρητήρια και συγχαρητήρια και για το διορισμό σας. Δεν ξέρω αν έχουμε συναντηθεί και προηγουμένως, όμως είμαι ένας έντρεμο οπαδό της Λατινικής Αμερικής. Δεν έχουμε Πορτογάλους και Ισπανούς ε, βουλευτές βέβαια ακόμα, αλλά αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα και η αποστέρησή τους είναι ένα σημαντικό θέμα. Όσα έγιναν από τον Κάστρο εμέσως ή άμεσα και εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές, ελπίδες για αλλαγές στο πολίτευμα, δεν θα υπάρξει και αλλαγή. Όμως πάντοτε επιθυμούμε η Κούβα να αλλάξει και να βελτιωθεί το ίδιο ε, και για την Ονδούρα και τη Βενεζουέλα. Όμως η εξισορρόπηση είναι ότι υπάρχουν γεωπολιτικές απειλές στην άμεση γειτονιά μας, στην δίπλα πόρτα με όσα συμβαίνουν με τη Ρωσία ή με τις παρεμβάσεις της Κίνας κάποιες φορές. Οπότε είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο να σκεφτούν το τι συμβαίνει και κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μια θερμάση των σχέσεων με την Λατινική Αμερική και να βελτιώσουμε τι γεωπολιτικές μα σχέσει σε διμερέ αλλά και πολυμερέ επίπεδο. Θα ήθελα, αν, αν μπορείτε, να σχολιάσετε το ευρύτερο τοπίο του ε, τι θα γίνει στην επόμενη θητεία και επειδή θα αναλάβει την ναύτα και την TTIP και τις εξετάσεις, την εξετασή του στο το, η επόμενη Το τι θα γίνει λοιπόν από την πλευρά της Χιλής και την επέκταση του διατλαντικού εμπορίου προς την Ασία. Εσείς βλέπετε την επόμενη 20 ετία να υπάρχει ένας τεράστιος χώρος ε, κοινών ιδεών, αρχών ε, και εμπορικών σχέσεων περνώντα από την Ιαπωνία μέσω της Λατινικής Αμερικής ως την Ευρώπη. Μήπως πρέπει να κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση αντί να κοιτάμε προς Ανατολές. Ευχαριστούμε η κυρία Λέζινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και πολύ για την παρουσίαση αυτή. Θα είμαι σύντομη, θα ήθελα εδώ απλά να εκφράσω το εξής από πλευράς της ομάδας μου. Αυτό το βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια διημερή συμφωνία σύνδεσης και συνεργασίας με την Κούβα είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε. Ελπίζουμε διαπραγματεύσεις μέσω πολιτικού διαλόγου να εξελιχθούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία συνεργασίας, να γίνουν διαπραγματεύσεις με αμοιβαίο σεβασμό, να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Κούβας. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι είναι το μοναδικό κράτος της, του κόσμου με το οποίο έχει τόσο ιδιαίτερη σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία άλλη χώρα, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση, από την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, η διαμόρφωση ενός κανονικού καθεστώτος με την ε, Κούβα θα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σημαντικό θα ήταν επίσης να έρθουν και τα ειδικά ε, μέτρα. Ευχαριστώ πολύ κύριος Κράσλερ Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Το παιχνίδι με την Κούβα δεν έχει τέρμα προχωρήσαμε μετά το 2000, έγινε ένα βήμα προς τα πίσω. Έγιναν προσεγγίσεις, έγιναν κάποιες δηλώσεις τις οποίες δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις, η αδερφή Κάστρο, το καθεστώς θα πρέπει να αλλάξει και πρόκειται να αλλάξει. Το διαπιστώσαμε αυτό στις επισκέψεις μας. Αυτό που δεν θέλει ο λαός της Κούβας είναι αυτό να έρθει από, έξι, από έξω. Να τους ε, προδιαγραφεί αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Είναι πάρα πολύ περήφανοι, όπως και οι Ισπανοί. Δεν θα ρίνουμε από οικοκρατικές συμπεριφερώσεις. Και αυτό το βλέπουμε και στην Αργεντινή και αλλού. Το Μάρτιο θα έχουν κλείσει 50 χρόνια από το πραξικόπημα στη Βραζιλία. Δεν υπήρχε τότε και με αυτή τη μορφή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ακολουθήθηκαν λοιπόν διπλά μέτρα και σταθμά, αναπτύχθηκε βιομηχανία και δεν μας ένιωσε τίποτα. Εδώ στο Κοινοβούλιο πάντα διατηρούμε διπλά μέτρα και σταθμά. Με την Κίνα δεν ξέρουμε τι να πρωτοπρολάβουμε και στην Κούβα τι κάνουμε. Στη Ρωσία είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί. Αν υπάρξουν κυρώσεις, λέμε καταρχάς οι γερμανικές επιχειρήσεις και όχι οι ισπανικές ή οι πορτογαλικές. Αρκεί να μην υπάρχει μεγάλο κόστος. Θα συνεχίσουμε, θα καταλήξουμε κάπου με την Κούβα. Αυτό είναι το βασικό. Και πώς ε, επηρεάζεται η κατάσταση από την Βραζιλία. Και όταν συζητάμε θέματα ε, για την Κρυμαία, να θυμηθούμε και το 1962 όταν υπήρχε αυτό το σχέδιο η κατάσταση πυράβλων στην Κούβα. Τότε κανείς δεν βγήκε να πει ότι θα διακηρύξουμε, θα ξεκινήσουμε πόλεμο με την Κούβα. Θα συμφωνήσουμε ποτέ. Έχουμε και μεγάλα προβλήματα με την Κριστίνα και στην Αργεντινή. Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με στην Μερκοσούρ. Αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο. Ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος, αλλά θα πρέπει και από τις δύο πλευρές να υπάρχει αποτέλεσμα. Και μου μένει και πέντε δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για τα σχόλιά τους. Ίσως να ξεκινήσω από αυτό που ονόμασε ο κύριος Τάνοκ την ε, ευρύτερη εικόνα, το ευρύτερο τοπίο και μετά να προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε λεπτομέρειες. Δεν είμαι συμπατριώτη σα, παρόλο που ε, πέρασα πολύ χρόνο στην χώρα σα ε, και έχω χάσει βέβαια και την προφορά του Κάρντιχ που είχα. Δυστυχώ. Αλλά νομίζω είναι λογικό να πει κανεί, αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινεί, κοιτάζοντα ανά τον κόσμο τι συμβαίνει, ότι οι χώρε του δυτικού ημισφαιρίου την Νότιο, την Κεντρική και την ε, Βόρεια Αμερική, μάλλον είναι οι χώρες με τις οποίες έχουμε το μεγαλύτερο βαθμό κοινών χαρακτηριστικών στην θεώρηση της κοινωνίας όπως την αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή την αντίληψή μας περί κοινωνίας, τι μορφή θα πρέπει να έχει και τις σχέσεις μεταξύ κοινωνίας των επίσημων δομών της κοινωνίας και των ατόμων. Όλα αυτά βάσει κοινή ιστορίας, γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού, αλλά και της αξιοσημείωτης πρόοδου που έχει γίνει σχεδόν σε όλη τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν διαφορετικές τάξεις τάσεις αλλά είναι δημοκρατικά τα καθεστώτα και αρκετά έντονη η ζωή τους από τότε που οι ε, χώρες αυτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Εξιοσημείωτη λοιπόν πρόοδος προς, προς την ανοιχτή τη συμμετοχική διακυβέρνηση. Το ευρύτερο το οποίο λοιπόν νομίζω μπορεί να μας ε, επιτρέψει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες προκλήσεις στην εδραίωση αυτής της πρόοδου. Δηλαδή, να περάσει κανείς από την επίσημη δημοκρατία στην αποτελεσματική και λογοδοτούσα και ανοιχτή εκπροσώπηση, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το να κερδίσει κανείς εκλογές ε, ανά πενταετία δεν είναι ακριβώς το σταθερότερο πρότυπο το οποίο επιζητούμε εμείς. Και βεβαίω πρότυπο δεν είναι όλο και περισσότεροι Λατινοαμερικάνοι πολίτε, οι Λατινοαμερικανικέ κυβερνήσει ε, να εναλλάσσονται κατά αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε και άλλε ευκαιρίε για διάλογο και άλλε ευκαιρίε για συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Δυτικού Ημισφαιρίου. Το διάλογο λοιπόν αυτόν τον έχουμε ξεκινήσει και υπάρχουν και άλλοι τομείς συνεργασία που επιδιώκουμε να ανοίξουν. Αυτό το πράττουμε με φιλοδοξία. Και πιστεύω και με ολοένα εντυνόμενη εμπιστοσύνη, με σχέσεις εμπιστοσύνης με τις περισσότερες χώρες. Μόλις ε, ήρθα στην ε, συνεδρίαση αυτή, επιστρέφοντας, από την ε, πιο πρόσφατη ε, συνάντηση για το διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε μια φανταστική διαδρομή τα τελευταία δύο χρόνια από ένα βαθμό αμυντικής επιφυλακτικότητας από τη μεξικανική πλευρά και μεγάλη, μεγάλη επιφύλαξη να ξεκινήσουν συζητήσεις με την κοινωνία των πολιτών προς μια πάρα πολύ φιλόδοξη ατζέντα, μεγάλο βαθμό αυτοκριτικής, πολλές επίμονες ερωτήσεις για αναζήτηση νέων τομέων συνεργασίας και ενεργό αναζήτηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτό μέσα σε μόλις λίγα χρόνια ανάπτυξης αυτού του διαλόγου. Μπορώ να σας δώσω πολλά παρόμοια παραδείγματα. Νομίζω λοιπόν ότι η ευρύτερη εικόνα μας επιτρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τη θέση που έχουμε καταλάβει και να επιδιώξουμε την ατζέντα που έχουμε καθορίσει με όλους τους εταίρους μας στο δυτικό ημισφαίριο. Από τον Καναδά στα βόρεια μέχρι την Αργεντινή και τη Χιλή στα νότια. Σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχουν δυσκολίες και σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι βραδία η επίτευξη αποτελεσμάτων όπως τις διαπραγματεύσεις με την Κούβα. Όμως είμαι βέβαιος ότι και εκείνοι στο συνολικότερο τοπίο μπορούν να προχωρήσουν και εμείς πιστεύω ότι μπορούμε και θα το παίξουμε, μπορούμε να επιτελέσουμε πρόοδο. Τώρα, για να απαντήσω στον κύριο Σαλαφράγκα, είναι δύσκολο για μένα να σας ορίσω ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων με την Κούβα. Είμαστε μόλις στα πρώτα βήματα και ήταν πολύ μεγάλη μου ικανοποίηση που μπορούσα να έρθω να σας πω σήμερα ότι θα υπάρξει έναρξη διαλόγου σύντομα. Χθε βέβαια μόλι το βράδυ έμαθα ότι για τον κουβανό ομολογό μου δεν ε, βολεύει η ημερομηνία που είχαμε προκαθορίσει. Αλλά δεν είναι παιχνίδια τακτική ούτε ελιγμή αυτά από πλευρά μα. Μόλι οριστεί η σωστή ημερομηνία ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε μάλλον με το ρυθμό ε, ε, ενός γύρου επίσημων διαπραγματεύσεων μία φορά ένα δίμηνο και με πολλές άτυπες συνομιλίες στο ενδιάμεσο. Το πώς βεβαίως θα προχωρήσουμε θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από την ε, κουβανική πλευρά. Το πώς θα αντιδράσουν στις προτεραιότητες που έχουμε καθορίσει. Γνωρίζουν ότι οδήποτε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλάβει τις συνήθεις διατάξεις που αφορούν τη διακυβέρνηση, το δημοκρατικό καθεστώς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, έχουν επιβεβαιώσει ατύπως ότι δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα όλο αυτό. Και ως συνήθως φαντάζομαι ότι τις πραγματικές δυσκολίες θα τις αντιμετωπίσουμε στις λεπτομέρειες, αλλά επί της αρχής συμφωνούν. Γνωρίζουν ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι διπραγματεύσεις με την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ακόμη σε ισχύ. Δεν μπορώ όμως να τους δώσω ούτε προβλέψεις, ούτε βεβαιότητα για το πότε αυτή η κοινή θέση θα πάψει να ισχύει η ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών στο Συμβούλιο ε, έφερε σε ισχύ την κοινή αυτή θέση και μόνο έτσι μπορεί και να αρθεί η ισχύ τη. Συμφωνούμε όμως με τους κουβανούς μας ομολόγους ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν ασχέτως αυτής της κοινή θέση. Θα έχουμε υπόψη και έχοντας υπόψη βέβαια πάντοτε το περιεχόμενό της οι με το Εκουαδόρ. Είναι τρόπον την πιο ε, άμεσες διότι ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα λίγο πολύ. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που περίπου που έχει ήδη περιληφθεί στις συμφωνίες με, ε, με το Περού και την Κολομβία. Υπάρχει δηλαδή ένα προκαθορισμένο πλαίσιο για τι δημοτεύσει με το Εκουαδόρ. Βεβαίω θα προσαρμοστεί στι ε, ιδιαιτερότητε τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά το πεδίο αυτών των αλλαγών θα είναι αρκετά, αρκετά μικρό. Δεν είναι μια χώρα που να διαφέρει τόσο αισθητά από του δύο γειτονέ τη, στα βόρεια και νότια, οπότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τους συμπεριλάβουμε τα θέματα των επενδύσεων παραμένουν ένα ζήτημα ανησυχία. Οι ε, εκπρόσωποι του Εκουαδόρ το γνωρίζουν και τις τελευταίες ε, εβδομάδες έχουν κάπως ε, μετριάσει την, τις διατυπώσεις που χρησιμοποιούν, τις έχουν κάνει πιο μετριοπαθείς, δίνοντας περισσότερες εγγύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη κυρίως ως προς το επίπεδο προστασίας. Λένε ότι αυτό δεν θα υποβαθμιστεί σε σχέση με τις ισχύουσες διμερείς συνθήκες. Αυτό λοιπόν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη και θα παραμείνει ένα καθοριστικό στοιχείο της συνολικής μας προσέγγισης για τις διαπραγματεύσεις με τη Μαρκοσούρ. Θα ήθελα να μπορώ και εδώ να σας δώσω μια ακριβή ημερομηνία, και ίσως να είμαστε σε, καλύτερα, σε, θέση να το κάνουμε αυτό περισσότερο μετά την Παρασκευή. των θα συναντηθούν οι διαπραγματευτές για τα εμπορικά ζητήματα. Θα δούμε τότε αν έχουμε αρκετή ουσία. Οι ενδείξεις που έχουμε λάβει δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα, ότι τις ε, διευκρινήσεις αυτές τις έχουμε λάβει μεμονωμένα από τα κράτη-μέλη της Μερκοσούρ. Εάν τις ε, συνδυάσει κανείς σε μία νέα προσφορά, βλέπει κάποιες αντιφάσεις μεταξύ των ε, μεμονωμένων εθνικών προσφορών. Οπότε αυτό μειώνει το ύψος των φιλοδοξιών. Θα πρέπει οι χώρες της Μερκοσούρ να βεβαιωθούν ότι το επίπεδο των φιλοδοξιών τους θα παραμείνει υψηλά ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν μαζί μας εφόσον αυτό επιθυμούν. Για το Μεξικό και τη Χιλή δεν περιμένουμε την ε, TTIP. Πιστεύω ότι χρειάζεται παράλληλη δράση. Το γεγονό ότι διαπραγματευόμαστε με έναν εταίρο δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να, να διαλλαγούμε και με άλλον. Υπάρχουν βεβαίω κάποια όρια και κάποιοι εμπειρογνώμονε μπορούν να βρίσκονται σε μια αίθουσα συνομιλιών μόνο με έναν εταίρο κάθε φορά. Δεν είναι τη υπόστατη. Αλλά προχωρούμε και με το Μεξικό και με τη Χιλή. Η Χιλή και η κυβέρνησή της χρειάστηκε πολύ χρόνο για να μας κάνει αντιπροτάσεις σε σχέση με την αναβάθμιση της συμφωνίας και μετά την σύνοδο στο Σαντιάγκο την περσινή χρονιά. Είναι λιγότερο προχωρημένο το στάδιο των διπλωματεύσεων με τους Χιλιανούς από ότι με τους Μεξικάνους. Όμως ε, δεδομένης της προόδου που επιτελέσαμε με το Μεξικό, νομίζω ότι μόλις φτάσουμε στη σύνταξη διαπραγματευτικής, στην εντολής και μόλις έχουμε συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές και αρχίσουμε να συνομιλούμε με τους, Μεξι... με Μεξικανούς, όλοι οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις θα το γνωρίζουν και έτσι θα προχωρήσουμε γοργά προς το στόχο της αναβάθμισης της συμφωνίας. Ίσως ένα τελευταίο σχόλιο να επανέλθω ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κούβας αλλά και σε κάποιους άλλους από τους γύρους διαπραγματεύσεων. Δεν είμαι βέβαιος εάν θα μπορούσα να συμφωνήσω με όσους λένε ότι εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και διπλά σταθμά. Πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε να πετύχουμε ως προς τα πρότυπα σε κάθε, σε κάθε ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Αλλά το είπα και στην αρχική μου απόκριση ότι η ευρύτερη οικονομική και κοινωνική αντίληψη που είναι κοινή μεταξύ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής σημαίνει ότι και εμείς αλλά και οι εταίροι μας από τη Λατινική Αμερική έχουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών. Αλλά ακριβώς επειδή τέτοιες σχέσεις επιδιώκουμε θα πρέπει να προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι να φτάσουμε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Νομίζω ότι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να αποστείλουμε σε όλους μας τους εταίρους σε αυτή την γεωγραφική περιοχή είναι ακριβώς αυτό στους εταίρους με τους οποίους έχουμε διαπραγματεύσεις, συνομιλίες, αλλά ακόμη και σε αυτούς με τους οποίους δεν έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία. Όσους ζουν κάποιες δυσκολίες, έχουν δυσχέρειες αυτόν τον καιρό, όπως με τη Βενεζουέλα, με την οποία δεν έχουμε συμβατικές σχέσεις, αλλά είναι σημαντικό να τους δείξουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Μερκοσούρ, τι επίπεδο φιλοδοξιών ή επιδόσεων θα αναμέναμε από οποιονδήποτε εταίρο είναι μέλος της Μερκοσούρ. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν αυτές έχουν αντίκτυπο, πηγαίνουν πέραν του αυστηρού πλαισίου της κάθε σχέσης και νομίζω ότι μας βοηθούν να τονώσουμε το κύρος και την αξιοπιστία μας σε όλη αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να έχουμε συστηματικές ε, επαφές. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα και πόσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Βεβαίως, η Κούβα είναι μια εξαίρεση, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θα δούμε τι τροπή θα πάρουν και αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, I would like to announce that... Uh, θα ήθελα να σας αναγγείλω το επόμενο σημείο. Δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Στέφανο Μασερβίζη, προσφάτω διοριστέντα επικεφαλής αντιπροσωπής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Οπότε παρακαλώ να μείνετε όσοι δικαιούστε, αλλά όσοι δεν ε, επιτρέπεται να είστε παρόντες και κλεισμένο το θηρόν συνεδρίαση ε, να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Παραλαμβάνω, η συνεδρίαση από εδώ και πέρα θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.